θέσω περιβαλλοντική ένωση. Μία δεκαετία μετά την αρχή της, πολλοί από τους συμπολίτε μας εξακολουθούν να ε, υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κρίσης λόγω ε, ανισότητας στους μισθούς, ε, μείωσης των μισθών και επισφάλειας. Η κρίση αυτή συνέδεσε την Ευρώπη με την ιδέα της λιτότητας. Βεβαίως, ορισμένοι πάντα αντιμετώπιζαν λιτότητα γιατί ήταν φτωχοί. Αντιμετώπισαν όμω και αυτού οι οποίοι ποτέ δεν, ήταν, ε, δεν αντιμετώπιζαν λιτότητα και ήταν υπεύθυνοι για την ε, χρηματοπιστωτική κρίση που έθιξε όλε μα τι κοινωνίε. Το αποτέλεσμα ήταν, ήταν η ανισότητα. Ιδιαίτερα η ανισότητα μεταξύ γενεών, δηλαδή η ανισότητα των νέων, δηλαδή επιπλέον η ανισότητα των φίλων. Γιατί οι γυναίκες θίγονται πολύ περισσότερο, πολύ πιο έντονα από την ε, επισφάλεια και την ε, ανισότητα στην ε, ευημερία. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν ε, διαιρέσει στι κοινωνίε μα και μα διαίρεσε και εμά. Διαίρεσε τι χώρε του Νότου και τι χώρε του Βορρά, τη Ανατολή και τη βύση, του δανειστέ από του δανειζόμενου. Άρα πρέπει να κλείσουμε αυτή την φάση. Πρέπει να αποκτήσει νέα νομοποίηση η Ευρώπη μεταξύ των πολιτών τη. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να απαιτήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη των δικαιωμάτων. Η κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι ουσιώδης πυλώνας και είναι νομίζω παράδειγμα μοναδικό στον κόσμο τον, ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν τέτοια συνοχή. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση με την ευρωπαϊκή προστασία να είναι ευκαιρία και όχι απειλή. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή με σαφείς στόχους, μετρήσιμους για την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και για την βιωσιμότητα του κράτους κοινωνικής προνοίας. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτήν την ε, πλευρά στις ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές και στην πολιτική συνοχή. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πρότασης που ε, πρότεινε στο Συμβούλιο η Ισπανική Κυβέρνηση η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας. Ένα πραγματικό backstop για τους συμπολίτε μας ούτω ώστε να αποκτήσει περιεχόμενο η τόσο σημαντική έννοια της αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής ηθαγένεια. Είναι μια ιδέα που θα προτείνουμε παράλληλα με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε το καθήκον που μας ανέθεσαν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, την οδηγία συνδυασμού τη προσωπική και εργασιακή ζωή και την οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμες ε, συνθήκες εργασίας. Πρέπει να διαβεβαιωθούμε ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τη φυλή τους, το φίλο τους και την ηλικία τους, θα πρέπει να έχουν ε, αξιοπρεπή εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταπολεμήσει την επισφάλεια στην εργασία, την ε, ανασφάλεια, γιατί δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η ιδέα ότι οι νέοι θα ζήσουν χειρότερα από τι προηγούμενε γενιέ. Είναι θεμελιώδε και αυτή είναι η θέση τη Ισπανική κυβέρνηση. Να, να προωθηθεί η εγγύηση για του νέου. Κυρίε και κύριοι, πριν από 7 μήνε η Ισπανία ε, απέκτησε μια κυβέρνηση με τι περισσότερε γυναίκε από όλε τι ε, κυβερνήσει των χωρών ΩΣΑ. Είναι ένα ορόσημο σε μια πορεία που έχει ακόμη πολλά βήματα μπροστά τη. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την πορεία εάν δεν είχε δώσει την ιδέα και την έμπνευση η Ευρώπη. Σήμερα εδώ μέσα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάνουν οι γυναίκες βουλευτές όλης της Υπήρου ούτω ώστε να προωθηθεί ο ε, φεμινισμός που είναι μέρος του κοινωνικού κεκτημένου. Σήμερα σας διαβεβαιώ ότι η Ευρώπη δεν θα κάνει κανένα βήμα πίσω. Θα κάνει περισσότερα βήματα μπροστά. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια τη Ευρώπη. Γι' αυτό σήμερα προτείνω να εγκρίνουμε μια στρατηγική ισότητα φίλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με δεσμευτικό χαρακτήρα. Μια στρατηγική για να καταπολεμήσουμε το χάσμα μεταξύ των γενεών και την ε, μεγαλύτερη απασχόληση και επισφάλεια ε, που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Η φωνή της Ευρώπης να είναι επικεφαλής στον αγώνα για το να γίνει 21ο αιώνας αιώνας των γυναικών. Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικέ οι αρχέ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ισότητα ευκαιριών για την πρόσβαση στην αγορά εργασία και σωστέ συνθήκε εργασία και η προστασία και η κοινωνική συμπερίληψη των πάντων. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό βασίζομαι στον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Αρχή ε, για την Εργασία για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στον αγορά εργασία. Ευρώπη θα πρέπει να ξέρει να δώσει περισσότερε ίσε ευκαιρίε και να τι εγγυάται στην πρόσβαση σε όλε τι μορφέ μόρφωση, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, στον πολιτισμό, στην ε, επιστήμη, στην έρευνα. Συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε ένα προπύργιο ουσιώδες έναντι εκείνων που θέλουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό όνειρο. Κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε εγγυήσει για την ασφάλεια των πολιτών μας και να ενισχύσουμε το ρόλο μας στον κόσμο, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στην Ευρώπη της ασφάλειας και στην Ευρώπη της άμυνας. Εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσαμε την μόνιμη διαρθρωτική συνεργασία για να δημιουργήσουμε ικανότητες στον τομέα της άμυνας μετά από δεκαετίες παράλυσης Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις τώρα, να προχωρήσουμε ξεκάθαρα στη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι είναι μια soft power εξ επιλογής και όχι εξ αδυναμίας. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το ρόλο μας και πέραν των συνόρων μας και η πολιτική βούληση για να το πετύχουμε αυτό είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση του ρόλου μας διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ελκυστικό πρότυπο για τον κόσμο σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι ακριβώς η Ένωση που θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Εκπροσωπούμε τις δυνατότητες που παρέχει η πολυμερής συνεργασία και η πολυμερής διεθνής τάξης που βασίζεται στο δίκαιο και στους ε, ε, κοινά αποδεκτούς κανόνες. Η Ισπανία, πρέπει να το πω αυτό, θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου λόγω και των ε, <clears throat> ειδικών σχέσεων που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και το βάρος της Ευρώπης είναι πολύ κατώτερο από αυτό που θα της άξιζε και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να είμαστε ένας πραγματικός παγκόσμιος εταίρος. Για να το πετύχουμε πρέπει να καταργήσουμε τον κανόνα της ομοφωνίας, όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και σε θέματα φορολογίας, σε θέματα πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού και στα θέματα του ελέγχου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη λοιπόν και να της δώσουμε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ευέλικτες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, τη νέα αυτή κυριαρχία. Τρίτον, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αρχιτεκτονική του ενημέου νομίσματος και να προχωρήσουμε στα πλαίσια του πολιετούς οικονομικού προγραμματισμού. Εδώ και 50 χρόνια στην Χάγη οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας των κρατών μελών και των κυβερνήσεων της Οικονομικής τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τη διαδικασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και από τότε ε, κάθε δεκαετία, στο τέλος κάθε δεκαετίας υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το 69 η κορυφή της Χάγης, το 79 το ενιαίο νομισματικό σύστημα, το 89 το σχέδιο Ντελόρ, και το 1999 η ίδρυση επίσημα του ευρώ. Βέβαια το κενό του 2009 δείχνει ακριβώς ε, τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν όταν η διεθνής δημοσιονομική κρίση απέδειξε και έφερε στην επικαιρότητα τις αδυναμίες της αρχιτεκτονικής ε, του ευρώ. Έτσι μπορούμε να δούμε καλύτερα τις επιπτώσεις της κρίσης ε, λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης θετικού συμβάντος το 2009. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το 2019 ε, και πρέπει να πούμε ταυτόχρονα ότι το ευρώ είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια που ωφελεί οικονομικά και πολιτικά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις γιατί αλλιώς θα μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ατελής και εκτεθειμένη στην αστάθεια. Το θέμα δεν είναι να ενισχύσουμε μόνο το δημοσιονομικό σύστημα, αλλά να μπορέσουμε μέσω της Τραπεζικής Ένωσης να προχωρήσουμε ε, <clears throat> στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων εφόσον υπάρξουν κρίσεις στο μέλλον. Ε, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε η Ευρώπη να ανακτήσει το ρόλο της σε αυτόν τον τομέα και οι πολίτες θα πρέπει να είναι ε, γνώστες αυτών, πρωταγωνιστές αυτών των μεταρρυθμίσεων που θα προστατεύσει τις καταθέσεις τους, θα τους προστατεύσει από τον πληθωρισμό και από τις κειμενόμενες οικονομικές κρίσεις. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα βοηθήσει και να προχωρήσουμε σε επίπεδο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή είναι η σωστή στιγμή όταν έχουμε συγκεκριμένες ευνοϊκές οικονομικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε τις οικονομικές αλλαγές. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε τη δομή του ευρώ πριν από την επόμενη κρίση η οποία μπορεί να αποδυναμώσει το νόμισμά μας και την ένωσή μας. Μαθαίνουμε από τις εμπειρίες που είχαμε μέχρι τώρα και προχωράμε με αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς. Αυτό είναι απαραίτητο και για τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά κυρίως για τους, αυτούς τους οποίους ε, εκπροσωπούμε τους ίδιους τους πολίτες. Σχετικά με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, νομίζω ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε στρατηγικές πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική και οι πολιτικές συνοχής πολύ σημαντικές για χώρες όπως η Ισπανία. Οι αστικές περιοχές δεν θα πρέπει να απομακρυνθούν από την Ευρώπη της υπαίθρου. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν μειώσουμε τον προϋπολογισμό θα δεχθούμε μια Ευρώπη της οποίας θα μειούται συνεχώς η σημασία. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί σαν μήνυμα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ικανοποιεί την ε, Ισπανική κυβέρνηση γιατί έχει καλά στοιχεία όπως η εξωτερική πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική, το επίπεδο των δαπανών, η ενίσχυση κάποιων προγραμμάτων καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη. Πρέπει η Ευρώπη φυσικά να είναι κυρίαρχη στον τομέα της καινοτομίας και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, της κβαντικής πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας και του αυτοματισμού. Μόνο όταν προχωρήσουμε τότε θα υποστηρίξουμε σωστά και τις προτάσεις για, την για τον διπλασιασμό του προγράμματος Εράσμους. Υπάρχουν φαινόμενα λοιπόν τα οποία οδηγούν δυστυχώς στην αύξηση της ανισότητας και στην παιδική ένδια. Νομίζω ότι η Ευρώπη των ευκαιριών, η πραγματικά καλή για τους πολίτες Ευρώπη ξεκινάει από την παιδική ηλικία και γι' αυτό ακριβώς η εγγύηση για την παιδική ηλικία είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την καταπολέμηση του αποκλεισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού. Κυρίε και κύριοι, η πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας έχει κάποια κενά, αλλά είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης και πρέπει όμως να υπάρξει ένα άλμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει πολύ περισσότερο από το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Πρέπει να είμαστε σωστοί στις δαπάνες, πρέπει να ικανοποιήσουμε όμως και τις προτεραιότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τα δίκτυα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Θέλουμε έναν προϋπολογισμό λογικό, προληπτικό, ο οποίος να δημιουργεί ευκαιρίες, να δημιουργεί συνέργειες και εξοικονομήσεις κλίμακας. Έτσι θα προχωρήσουμε στην προστασία της Ευρώπης, μια Ευρώπη κοινωνική, μια Ευρώπη άμυνας, μια Ευρώπη οικονομική και νομισματική. Θα πρέπει εμείς να έχουμε ένα σωστό επίπεδο ανάμεσα στα μέσα και στους στόχους. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επανέλθω στην ιδέα να αντιμετω... για την τελευταία για το τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής μου σε σχέση με θέματα όπως οι προκλήσεις στις κλιματικές αλλαγές και στη μετανάστευση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να βασιστούμε στις ευρωπαϊκές αρχές. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά σύνορα. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες και σε συνενέσεις που ε, θα ξεπεράσουν τις διαιρέσεις. Βέβαια η τομείς αυτή είναι το πεδίο μάχης για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν θα πιστέψουν ποτέ στην Ευρώπη. Είναι το χαρακτηριστικό αν θέλετε κομμάτι αυτών που θέλουν να υπονομεύσουν την φιλελεύθερη δημοκρατία. Και για μια ακόμη φορά το σημαντικό είναι να προστατεύσουμε την Ευρώπη, να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών, στα διεθνή φόρα ακούγονται όλο και περισσότερο κάποιες θέσεις σκεπτικιστικές για να μην πω ξεκάθαρα πολεμικές. Η προοπτική μας στο πλαίσιο αυτό είναι να οδηγηθούμε σε μια συμβιβαστική πρόταση που να ανοίγει ευκαιρίες για το μέλλον. Η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και της δικής μας χώρας. Τα ενεργειακά δίκτυα και οι διασυνδέσεις θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας και θα μειώσουν τις εκπομπές. Νομίζω ότι οι συνέπειες αυτών των προκλήσεων αν δεν αντιμετωπιστούν θα είναι καταστροφικές. Νομίζω ότι θα πρέπει και σε επίπεδο πολιτικής ένωσης να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε ο αυταρχισμός και ο υπερβολικός εθνικισμός που αποκλείει από την ανάπτυξη κομμάτια του πληθυσμού να μην μπορέσουν να οδηγήσουν σε έναν αρνητισμό ο οποίος δεν θα είναι τεκμηριωμένος φυσικά. Εμείς λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολλά σαν μια Ευρώπη η οποία θα συνεργαστεί και με τους υπόλοιπους σημαντικούς εταίρους σε διεθνές επίπεδο. Με τους ίδιους θόρους θέλω να αναφερθώ στο δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα το μεταναστευτικό. Μιλάμε για ένα θέμα κυρίες και κύριοι όπου η συνεργασία και ο συντονισμός και με τις χώρες προέλευσης και με τις χώρες τράνζιτ και με τις χώρες κατάληξης είναι σημαντικός και για την Ισπανία φυσικά αυτό είναι σημαντικό. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε, ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έγγραφο που προήλθε ε, από την συνεργασία με το Βασίλειο του Μαρόκου στον τομέα της συνεργασίας και ελέγχου. Εδώ έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο και πρέπει να το θυμίσω εμείς απαιτείται να κάνουμε μια νέα προσπάθεια στον τομέα αυτό. Η διάσκεψη του Μαρακές αντιπροσωπεύει, αντιπροσώπευσε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση την πολυμερή της μεταναστευτικής πρόκλησης και η Ισπανία είναι ένας από τους πρώτους που επικύρωσε την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στις κοινωνίες μας σε επίπεδο συζητήσεων θα πρέπει ε, να μην γίνεται συζήτηση αποκλειστικά για την παράνομη μετανάστευση, γιατί η τακτική, η νόμιμη μετανάστευση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Σε μία ήπειρο ε, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζεται από την γύρανση του πληθυσμού αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν συνεννοηθούμε με μια άλλη ήπειρο, την Αφρική, η οποία απαιτείται να περάσει από μια κοινωνικο-οικονομική βαθιά αλλαγή. Αυτός ο πολιτικός δρόμος, ο οποίος έχει μέλλον, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίος χώρος χωρίς εξωτερικά σύνορα έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά μια κεντρική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να μεταρρυθμιστεί το ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου και θα πρέπει οι δύο αρχές που θα χαρακτηρίσουν τη δράση μας να είναι η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη. Ε, προφανώς ε, είναι περίπλοκες οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, που κινδυνεύουν, θα πρέπει να σεβαστούμε και την νομική τάξη της κάθε χώρας. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές φορές βέβαια δράσει οι οποίες είναι αντίθετες μερικές φορές με τις βασικές ανθρωπιστικές αρχές. Ε, η Ευρώπη δεν πρέπει να ακολουθεί τις μόδες. Η Ευρώπη έχει ένα δημοκρατικό παρελθόν και δημιουργεί τις μόδες. Αυτή είναι και η δύναμή μας και η ισχύ μας. Κύριε βουλευτέ, ε, η μεγαλύτερη αδυναμία μα εδώ στην Ένωση είναι οι διαιρέσει μα που όπω είπα στην αρχή, εκείνοι που θέλουν να αποτύχει το μοντέλο μας. Ένα μοντέλο που βασίζεται σε ένα ε, το κύκλο. Η δημοκρατία, η πρόοδο και το κράτος ευημερία. Η υπέρβαση των αδυναμιών μα και των διαιρέσεών μα πρέπει να βασιστεί στην καταπολέμηση των, ε, αυτών των ε, στερεοτύπων. Το Μάη φέτος θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση. Ε, έχουμε απέναντί μας ένα μήνυμα που έκανε την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, πριν από λίγες δεκαετίες, ένα πεδίο μαχών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τα δικά μας ιδανικά τις προσπάθειες αυτές. Ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Το είδα με τα μάτια μου όταν ήμουνα στη δεκαετία του 90 στη Βοσνία εργαζόμενος για, την ε, για τα Ηνωμένα Έθνη σε μια πόλη που καταστράφηκε από, την, ε, από τον εμφύλιο πόλεμο και το μίσο στο Σαράγεβο. Η βαρβαρή, η βαρβαρότητα που θεωρούσαμε ότι είχε αποκλειστεί πλέον από την Ήπειρό μα ξαναεμφανίστηκε και τροφοδοτείται από δυνάμεις που πάντα ε, αντιπαραθέτουν το μίσος στην συμβίωση δεν απειλούν μόνο την προσπάθεια ενοποίησής μας. Με ε, έμεσο και, και ε, ύπουλο τρόπο αξιοποιούν ε, τα θέματα ορισμένων που λένε ότι είναι αντίθετοι σε αυτές. Ε, παρακαλώ λοιπόν το σώμα σας να μην επηρεάζεται από αυτούς. Απευθύνομαι σε εσά για να είστε αποφασιστικοί στην προστασία των ευρωπαϊκών αξιών. Και χρειάζεται δύναμη για να αντιμετωπίσετε τις ειρήνες του αυταρχισμού. Γιατί έχουν ένα μόνο στόχο. Στόχος είναι να καταστρέψουν την Ευρώπη. <clears throat> Γι' αυτό κάνω έκκληση σήμερα. Υπάρχει αναγκαιότητα να προστατεύσουμε την Ευρώπη, ούτω ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει του πολίτε τη τα επόμενα χρόνια. Είμαι πεπισμένο ότι θα προχωρήσει το κοινό μα εγχείρημα παρά τι δυσχέρειε. Θα έχουμε διαφορέ απόψεων, θα έχουμε ε, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι συνολικά θα έχουμε περισσότερη πρόοδο από οπισθοχωρήσει. Βεβαίως, ε, η πρόοδη αυτή δεν θα βρίσκει τους πάντες σύμφωνους, γιατί αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε, διότι οι ιδέες μας μπορεί να είναι διαφορετικές, μπορεί και αντιτιθέμενες, αλλά πρέπει να υπάρχει ε, προσπάθεια να συνδυαστούν αυτές οι ιδέες για να προχωρήσουμε διατηρώντας ε, την ευημερία μας σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Ούτως ή άλλως, παρά τις δυσχέρειες, έχουμε μια σταθερή βάση, την αλληλεγγύη στην πράξη, που αυξάνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε κάθε φορά που δυστυχώς υπέστημεν τρομοκρατικά χτυπήματα. Είναι, είναι ε, το σπέρμα μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όταν ένας Ισπανός πολίτης ε, σε αλληλεγγύη με μια τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι βάζει στο, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωση μια γαλλική σημαία αγκαλιάζει την ιδέα της Ευρώπης. Και όταν ένας Γερμανός ε, κάνει το ίδιο για την επίθεση στην Βαρκελόνη, αγκαλιάζει την ιδέα της Ευρώπης. Εδώ ξέρουμε ότι υπήρξε μια φρικαλαία επίθεση της, ε, στο Στρασβούργο πριν από ένα μήνα. Όταν εκφράζουμε όλη την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα, αγκαλιάζουμε τη σημαία της Ευρώπης. Οι εχθροί της Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ε, έναντι αυτού του αυξανόμενου αισθήματο ε, αόρατη αλλά πραγματική αλληλεγγύη και η οποία εκφράζεται κυρίω μεταξύ των πιο νέων προβάλλουν την ιδέα της Ευρώπης ως σύμβολο κατά της ανισότητας, κατά της αδικίας, κατά του αυταρχισμού, κατά της φαλοκρατίας, κατά του ρατσισμού ή για να εκφράσουν απλώς την ε, ε, ε, διαφωνία τους με αποφάσεις που είναι αντίθετες με τη λογική των καιρών και τα συμφέροντά τους. η... Το να ξεχάσουμε την ιστορία είναι μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Δεν μπορούμε να είμαστε διστακτικοί έναντι των αβεβαιοτήτων. Η αποφασιστικότητα θα μας επιτρέψει να επανακτήσουμε το ρυθμό μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα αυταρχισμό που ζει από μια επινοημένη νοσταλγία. Δεν υπάρχει χειρότερη νοσταλγία από το νοσταλγούμε κάτι που ποτέ δεν υπήρξε. Όπως λέει μια, ένα τραγούδι ενός μεγάλου Ισπανού τραγουδιστή. Σε όλε αυτές τι επινοημένε ε, νοσταλγίες ερωτώ. Είχαμε σταθερή ειρήνη όταν υπήρχαν ε, κλειστά σύνορα. Υπήρχε οικονομική πρόοδος όταν ε, τα τελωνία περιόριζαν ε, τις ε, συναλλαγές. Είχαμε περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα σε κάθε κράτος όπως τα έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια στα κράτη της Ένωσης. Πολύ κοντά σε εδώ, στα πεδία μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουμε την απάντησή μας. Γι' αυτό σήμερα θέλω να πω ότι έναντι της εσωστρέφειας πρόοδος, έναντι της ρητορική των ε, ε, αποκλειουμένων ταυτοτήτων, θέλουμε ταυτότητες που ε, συμπεριλαμβάνουν τους πάντες. Όπως έλεγε ένα σύντροφος από το Ισπανικό, από την Ευρωπαϊκή Σοδημοκρατία, ο καταπληκτικός Φραντ Τίμερμαν, το παρελθόν ποτέ δεν θα είναι το μέλλον για τις κοινωνίες μας. Το παρελθόν είναι ένα... Ε, ένα χώρο που μαθαίνουμε από τι επιτυχίε και τα λάθη μα. Πρέπει να κινητοποιηθούμε για την Ευρώπη. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ε, αξίες που κάνουν το εγχείρημά μας ε, ε, μοναδικό στον κόσμο και το οποίο το ζηλεύουν πολύ στον κόσμο. Μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε αυτούς που απ' έξω αλλά και από μέσα προσπαθούν να καταστρέψουν τα ειδόδη μας. Και θέλουν να το κάνουν, να μην το ξεχνάμε, και θέλω να το υπογραμμίσω και να το θυμίσω. Θέλω να το κάνω για ένα μόνο λόγο. Λόγω των αξιών που υποστηρίζουμε. Που υποστηρίζει η Ένωση. Πρέπει λοιπόν εμεί να απαντήσουμε υποστηρίζοντα αυτέ τι αξίε. Σε αυτή την πορεία, κύριε Βουλευτέ, χρειαζόμαστε πεποίθηση και αποφασιστικότητα. Πρέπει να συνδυάσουμε τα ιδεώδη μα με την προσπάθεια πραγματιστικών λύσεων όπω κάνουμε τα τελευταία 60 χρόνια κοινή ζωή. Το καθήκον μα ω κληρονόμοι αυτή τη μεγάλη κληρονομιά είναι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε αυτό που κληρονομήσαμε για να το περάσουμε στι επόμενε γενιέ. Εάν μάθαμε κάτι είναι ότι σε συγκεκριμένε συγκυρίες της ιστορίας μας, όπως αυτήν, το να αντισταθούμε είναι πρόοδο. Σήμερα, στις γενιές που εσείς εκπροσωπείτε σε αυτό το κοινοβούλιο, ανταποκρίνεται ένα καθήκον, να προστατεύσουμε την Ευρώπη, ούτως ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει τους πολίτες της. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα σύμφωνα με το Catch the Eye. Κλείνω το κατάλογο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη εγγραφεί. Οπότε ζητώ από τους εκπροσώπους των ομάδων να τηρήσουν ε, το χρόνο που τους έχει ήδη κατανεμηθεί. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε όλους τους συναδέλφους αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε το χρόνο σας. Πρώτος ομιλητής είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φραντς Τίμερμανς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Σάντσες για την πολύ εμπνευσμένη ομιλία του και νομίζω ότι η μία ιδέα που ήθελε να μοιραστεί μαζί μας είναι ότι αν η Ευρώπη θέλει να προστατεύσει τους πολίτες της, εμείς οι πολιτικοί έχουμε συλλογική ευθύνη να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Μόνο μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. Και αυτοί που πολλούν την αυταπάτη ότι μπορεί κανείς να προστατεύσει τους πολίτες απομονώνοντας όσους είναι διαφορετικοί, οικοδομώντας τείχους και φράχτες, πολλώντας ένα ε, απατηλό όνειρο ε, εθνικισμού θα οδηγήσουν στην απογοήτευση, διότι δεν υπάρχει προστασία στον προτεξιονισμό απομόνωση υπάρχει στον απομονωτισμό και τα έθνη όταν μείνουν μόνα τους στην Ευρώπη δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πολλές προκλήσεις που μας προσφέρει ο κόσμος. Μόνο μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί να κάνει αυτό που απαιτούν οι πολίτες, δηλαδή να τους προστατεύσει και να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν το μέλλον τους ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι άνθρωποι. Ξέρω ότι η Ευρώπη ε, υπάρχει στις φλέβες του ε, Πέντρο Σαντσές, ε, ανήκει στην τελευταία γενιά που μεγάλωσε υπό τη δικτατορία, μια γενιά που μεγάλωσε με το όνειρο της ελευθερίας και η Ευρώπη, η Ισπανία τώρα πια έχει αναλάβει την σωστή της θέση στην καρδιά της Ευρώπης. Το μήνυμα που έχω σήμερα στην κυβέρνηση της Ισπανίας είναι το εξή. Κοιτώντα τα τελευταία 40 χρόνια, νομίζω ότι σωστά μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη έχει διαμορφώσει την Ευρώπη διότι αυτή ήταν η επιθυμία του ισπανικού λαού. Νομίζω όμως επίσης ότι θα πρέπει να πούμε ότι και η Ισπανία θα πρέπει να συνδιαμορφώσει την Ευρώπη. Χρησιμοποιήστε το δυναμικό σας για να διαμορφώσετε το κοινό μας μέλλον. Είσαστε ισχυροί, ανθεκτικοί και έχετε δείξει στην τρομερή αυτή κρίση που αντιμετώπισε ε, η Ισπανία πώς μπορείτε να ε, την ξεπεράσετε και πιο ισχυρή. Ναι, πράγματι είναι πολύ ε, υψηλή ακόμη η ανεργία. Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια όμως. Και νομίζω ότι η αποφασιστικά του ισπανικού λαού αποτελεί έπνευση για όλους μας ε, στην Ευρώπη. Επίσης, ο λαός ε, της Ισπανίας ε, συμμερίζεται τις αξίες ελευθερία, δημοκρατία, ευημερία. Αυτά είναι πολύτιμα πράγματα και δεν θα πρέπει ποτέ να τα θεωρήσουμε δεδομένα. Η Ισπανία έχει σημαντική θέση στην Ένωσή μας και η ευρωπαϊκή της ιστορία πάει πολύ πιο πίσω από το 1985. Ιδιαίτερα όσον αφορά το πόσα χρωστά η Ευρώπη στην αποφασιστικότητα και τι ιδέε ανθρώπων όπω είναι ο Σαλβαδόρ Ντε Μαδαριάγα που βοήθησε να οικοδομηθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την ιδέα τη ε, ελεύθερη και δημοκρατική Ισπανία. Και οι άνθρωποι που δεν εγκαταλείπουν τα ιδανικά του ούτε στι πιο σκοτεινέ μέρε είναι αυτοί που μπορούν να διαμορφήσουν με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον μα. Είδε ότι η ταυτότητά μας, ε, η επιτυχία μας ε, είναι συνδεδεμένη του ενός ε, με του άλλου. Τώρα, 40 χρόνια μετά το Σύνταγμα της Ισπανίας, ε, βρίσκεστε στην καρδιά μιας Ενωμένης Ευρώπης η ανάπτυξή σας είναι στο 2%. Η ανεργία ακόμη είναι πολύ υψηλή, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν και υπάρχουν πολλά θετικά μηνύματα στην οικονομία. Η οικονομία έχει ορθοποδήσει και πάλι και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό οφείλεται στο θάρρος και την αποφασιστικότητα των Ισπανών και την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Την αλληλεγγύη αυτή την ανταπέδωσε η Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ε, βοηθήθηκε από την Ευρώπη, αλλά έχει δείξει επανειλημμένα ότι ε, δείχνει καθημερινά την αλληλεγγύη τη με το υπόλοιπο τη Ευρώπη. Το βλέπουμε αυτό στο θέμα τη μετανάστευση. Η Ισπανία και η Μάλτα, ακόμη και σε πολύ δύσκολου καιρού, ε, επιδεικνύουν αλληλεγγύη απέναντι σε ανθρώπου που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. εσύ ήσουν ηγέτης, καλωσόρισες εσύ τους, ε, του ε, ε, τους ναυαγούς στο πλοίο Aquarius. Στο όνομα του ισπανικού λαού είπες ότι δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να πνιγούν. Αυτό είναι πραγματική πολιτική ηγεσία. Δεν επέλεξε τον εύκολο δρόμο, δεν έστρεψε αλλού το βλέμμα, δεν κατηγόρησε του ε, ε, πρόσφυγε, απλά ανέλαβε την ευθύνη για τη μοίρα του. Ε, οι εικόνες των πλοίων αυτών και οι διαιρέσεις που ε, ε, δημιούργησαν ε, ακόμη και οι λίγες αφήξεις στις ακτές μας έδειξαν τις δυσκολίες και τώρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το κοινό σύστημα ασύλου. Μόνο με μεταρρυθμίσεις θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη λύση. Μόνο η προστασία των συνόρων δεν αρκεί. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ασύλου που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στι θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίση, Πέδρο, να τονίσω αυτό που είπε για την Αφρική. Εάν υπάρχει μία ήπειρος που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης, αυτή η ήπειρος είναι η Αφρική. Κανείς άλλος στον κόσμο δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είναι η ε, αδερφή ήπειρός μας. Ε, απέχει πολύ λίγο από τις ακτές μας και εάν δεν αναλάβουμε κοινή ευθύνη, συλλογική ευθύνη για το μέλλον και των δύο υπήρων, τότε τα προβλήματα της Αφρικής ε, δεν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε μακριά από την Ευρώπη όσο υψηλούς φράχτες και να χτίσουμε. Χρειάζεται ένα μέλλον στο οποίο να μπορούν να πιστέψουν οι άνθρωποι της Αφρικής. Χρειαζόμαστε σταθερότητα στην Αφρική, ώστε και η Ευρώπη να είναι σταθερή και ελεύθερη στο μέλλον. Πέδρο, σε καλό να Οδηγήσει την Ευρώπη ώστε να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και αν βρίσκονται. Στον προϋπολογισμό μας θα έχουμε σχεδόν ε, τριπλάσια αύξηση, 33 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για τα θέματα μετανάστευσης. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, όχι μόνο επειδή για την Ισπανία, όχι μόνο επειδή έχετε επιδείξει το, τόση αλληλεγγύη, αλλά επειδή γνωρίζετε και ε, τις, ε, τρομε, επειδή έχετε δει τρομερές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της. Με 9 δισεκατομμύρια ευρώ θα στηρίξουμε και τη τον ε, ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης σε κάτι το οποίο θα προωθήσει, θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας. Ε, επίσης, ε, πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κινητοποιηθεί με το σχέδιο Juncker και έτσι έχουν βοηθηθεί περίπου 45.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είδαμε δημιουργία θέσεων εργασίας και στήριξη της κυκλικής οικονομίας ε, στην Ισπανία. Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζω την προσήλωση της χώρας σας στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ε, πρέπει και η Ισπανία και η Ευρώπη να εφαρμόσει αυτόν τον μετασχηματισμό και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να χαιρετήσω τον συνάδελφό μου που κάθεται εδώ δίπλα μου που έχει φροντίσει σε όλο τον κόσμο, ε, έχει καταβάλει προσπάθειες ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του Παρισιού. Νομίζω ότι έχει ηγηθεί παγκοσμίω στο θέμα αυτό και ε, του αξίζει η αναγνώρισή μας και η εκτίμησή μας. Το νέο πρόγραμμα InvestEU ε, έχει τη δυνατότητα ε, να κινητοποιήσει επιπλέον 650 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις ανάμεσα στο 2021 και το 2027. Επίσης, θα υπερδιπλασιαστεί η χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Erasmus και είχα τη χαρά να ε, εργαστώ και στο παρελθόν ε, με τον δημιουργό του ε, προγράμματος Εράσμους. Πραγματικά πρόκειται για πολύ ισχυρό πνεύμα. Ο Χουάν Μαρίν είναι ο άνθρωπος αυτός. Και έχω δει πολλούς ε, νέους ανθρώπους ε, των οποίων ε, οι γνώσεις και το ανοιχτό πνεύμα έχουν εντυπωσιάσει όλους μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε σύμφωνα να συμφωνήσουμε πάνω στο νέο προϋπολογισμό και βασίζομαι στην υποστήριξη του Πέντρο, των ομολόγων του και του Κοινοβουλίου για να το πετύχουμε αυτό. Θα ήθελα να τονίσω την αξία, την ποιότητα του θεματολογίου της Ισπανικής κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σχέδιο για να κλείσουμε την ψαλίδα αμοιβών ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να κλείσουμε την ψαλίδα στις ε, συντάξεις ε, που ανέρχεται σε 40% στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή, να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες της Ευρώπης. είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή τη στιγμή και βασίζομαι στην κυβέρνηση του Πέντρο για για να ε, το πετύχουμε αυτό. Γιατί δεν έχουμε δώσει τέλος στη βία ει βάρο των γυναικών. Είναι υποχρέωσή μας αυτό, είναι καθήκον μας. Και γιατί δεν ονοματίζουμε αυτούς που ε, εσφαλμένα επικαλούνται οικογενειακές αξίες ε, για να στερήσουν από τις ε, γυναίκες τα πλήρη δικαιώματα. Ε, δεν επιτρέπεται να δικαιολογούμε τη βία στο, σε ένα γάμο, στο οικογενειακό πλαίσιο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ισπανία και η ευρωπαϊκή της ιστορία αποτελούν υπόδειγμα για την Ευρώπη. Δείχνει τι σημαίνουν οι αξίες για τις οποίες μιλάμε και δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε με τη συνεργασία και με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ευρώπη προστατεύει, αλλά πρέπει και εμείς να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο πρώτος ομιλητής εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων είναι ο επικεφαλής του ΕΛΚ, ο κύριος Μάνφρετ Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε η παρουσία σας εδώ δίνει μια μεγάλη όθηση για το 2019, γιατί εσείς είστε φιλοευρωπαϊστής, ε, ξεκάθαρα δεσμευμένος σε ευρωπαϊκούς ε, στόχους. Γι' αυτό είναι θαυμάσιο που σας έχουμε εδώ. Η Ευρώπη σημαίνει για την Ισπανία ειρήνη και ευημερία. Η Ισπανία σημαίνει για την Ευρώπη ισχύ, φρέσκες ιδέες και ηγεσία. Γι' αυτό είναι πολύ καλό που σας έχουμε εδώ. Από την άλλη, είναι σημαντικό γιατί το 2019 είναι το έτος όπου θα εορτάσουμε τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπα... ευρωεκλογέ θα λάβουν χώρα. Και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σα όσον αφορά την υποστήριξη του Φραντ ε, Τίμερμαν ως σοσιαλιστή υποψηφίου. Είναι μια σαφή ένδειξη ότι πιστεύετε στη δημοκρατική ιδέα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το κρατήσετε ζωντανό, ε, ε, θα κρατήσετε ζωντανή αυτή την αρχή και μετά τις ευρωεκλογέ. Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, δυστυχώ θα πρέπει να μιλήσουμε και για εθνικισμό και ρατσισμό. Έχουμε τα χθεσινά αποτελέσματα των εκλογών. Ε, ε, ε, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι βρίσκονται στο ίδιο πλοίο σύμφωνα με το πνεύμα των ιδρυτικών πατέρων της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές αξίες βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι εξτρεμιστές δεν έχουν χρώμα. Εσείς είστε ένας φιλοευρωπαϊστής, αλλά η κυβέρνησή σας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την υποστήριξη των ε, ακραίων ε, αριστερών και των ε, εκείνων που είναι υπέρ της απόσχησης. Ο στόχος όμως της Ευρώπης είναι να υπάρξει σταθερότητα και, να... και ο Φραντς Τίμερμαν εξήρε την θετική εξέλιξη τη Ισπανική οικονομία ε, τα τελευταία έτη μετά την οικονομική κρίση. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε όλου, αυτό έγινε χάρη στι προσπάθειε τη κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχώη να δημιουργήσει προποθέσει για αυτή την ε, οικονομική επιτυχία τη Ισπανία. Και τώρα εσεί ε, θέλετε να πάρετε πίσω τι μεταρρυθμίσει τη αγορά εργασία που έκανε ο Μαριάνο Ραχώη. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν το εσφασμένο μήνυμα όσον αφορά τη δημιουργία ενό οικονομικού μέλλοντο για την Ισπανία Γι' αυτό προποθέτει να κάνει κανεί μεταρρυθμίσει. Ε, μεταρρυθμίσεις, συγγνώμη. Η Ευρώπη θέλει να αυξήσει τα έσοδα των εργαζομένων. Άρα λοιπόν παρακαλώ να διατηρήσετε τι μεταρρυθμίσει, μην ακούσετε του λαϊκιστέ. Δεύτερον, ε, σεβόμαστε πάρα πολύ την κυβέρνησή σας, έστω και αν δεν συμμεριζόμαστε τις ίδιες πολιτικές αξίες και ιδέες αλλά μα ανησυχεί το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας. Αυτή τη στιγμή δεν ε, πετύχατε μια επικοδομητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για το προπολογισμό που παρουσιάσετε. Ωστόσο, εκπροσωπείτε μια από τις μεγαλύτερε οικονομίες στην Ευρωζώνη και μια τέτοια μεγάλη οικονομία χωρίς ε, προπολογισμό ε, οδηγεί σε αστάθεια. Και αυτό ε, και με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αστάθεια στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τη μετανάστευση, εμεί στο ΕΛΚ έχουμε ξεκάθαρε προτεραιότητε. Ε, το σχέδιο Μάσαλ για την Αφρική ένα φιλόδοξο πλάνο επαναγκατάσταση των προσφύγων. Θέλουμε να βοηθήσουμε του πρόσφυγε από τη Συρία και άλλε περιοχέ. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι η παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να τερματιστεί. Θα πρέπει ε, να ε, καταστρέψουμε το, να πατάξουμε το απάνθρωπο μοντέλο παράνομη μετανάστευση των διακινητών. Και εδώ η Ισπανία φέρει ένα μερίδιο ευθύνη. Τα να περάσματα από την Ισπανία έχουν διπλασιαστεί ε, τον τελευταίο χρόνο. Ακούω πολύ συχνά το επιχείρημα ότι είναι δύσκολο να προστατευτούν τα σύνορα. Εγώ ε, πέρσι το καλοκαίρι πήγα στην άλλη πλευρά της Υπήρου, στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Και εκεί φτιάχτηκε ένας φράχτης ύψους ενός ε, μέτρου για 100 χιλιόμετρα. Και αυτό μας δείχνει ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να προστατευτούν τα σύνορα ε, και τέτοια μέτρα ε, όπως ε, τέτοιος φράχτης είναι αποτελεσματικά. Εάν θέλουμε να πατάξουμε τον εξτρεμισμό θα πρέπει να προστρέξουμε σε τέτοια μέτρα και αναμένουμε από την Ισπανία να προστατεύσει τα σύνορα όπως στην Χάουτα και στη Μελίγια. Στην Ισπανία ε, υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις αποσχεστικές στάσεις στην ε, Καταλωνία. Εμείς ε, ως ΕΛΚ στηρίζουμε την ενδευτική αικαιρότητα της Ισπανίας και στηρίζουμε την κυβέρνηση όσον αφορά την διατήρηση της ενότητας της Ισπανίας. Η Ευρώπη έχει κονδομηθεί επί της αρχής του κράτους ε, δικαίου, το ίδιο και η Ισπανία. Και αυτό έπραξε και η κυβέρνηση Ραχώ και εμείς θα σας υποστηρίξουμε εάν θέλετε να προσφέρει στις ίδιες αρχές. Η δική μου πολιτική ομάδα ε, υπερψήφισε ένα κομμουνιστή αντιπρόεδρο, αλλά δεν θέλαμε να υπερψηφίσουμε έναν ακροδεξιό υποψήφιο, γιατί θέλουμε να εγγυηθούμε οι εθνικιστές να μην έχουν λόγο για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Έχετε πολλά πράγματα να κάνετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας και να σας ευχαριστήσω και για την ε, ε, βούλησή σας Ρωσίας ε, ε, όσον αφορά τις φιλοευρωπαϊκές ε, αρχές στην Ευρώπη. Όχι εθνικισμοί, αλλά ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας. Τώρα ουρουλάτη in aula. Serve sempre il veterinario. Prossimo intervento è quello dell'onorevole. Ε, παρέμβαση του κυρίου Ούντο Μπούλμαν. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυβέρνησης, αγαπητέ Πέδρο, καλώς όρισες ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αγαπητέ Πέδρο. Dear I, cannot help. I cannot help. Again quoting you. Αγαπητέ Πέδρο, δεν μπορώ παρά να αναφέρω τα λόγια σου. Αν η Ευρώπη πρέπει να μας προστατεύει, Πρέπει εμείς να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Μακάρι να ήταν αυτό το σύνθημα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Μακάρι να ήταν αυτό το σύνθημα όλων των Ευρωπαίων ηγετών και να αποτελεί το ορόσημο ε, έναντι το οποίο θα πρέπει να μετρηθεί οποιοδήποτε ε, με πολιτικές ευθύνες στην Ευρώπη. Δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό και γι' αυτό και σε περιμέναμε με ανυπομονησία. Θέλαμε να σε ακούσουμε αυτή την εμπνευσμένη και παθιασμένη ιδέα της ε, δικαιοσύνης και της προόδου για την Ευρώπη μας. Δυστυχώ δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, συνάδελφε κύριε Βέμπερ, όπω το παρουσιάζετε. Όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο σκάφο, αλλά εάν θέλουμε να πατάξουμε τον εθνικισμό, αν θέλουμε να παρεμποδίσουμε ότι η Ευρώπη να μην γίνει το θύμα των ακροδεξιών, τότε θα πρέπει το σκάφος αυτό να έχει και μια κατεύθυνση πλεύσης, θα πρέπει να αναπτύξει ένα δυναμισμό και θα πρέπει να εμποδίσουμε την τελμάτωση των, τις τελευταίες δεκαετίες όπου οι άνθρωποι στην Ευρώπη περιμένουν να παράσχουμε αποτελέσματα και να τις προστατεύσουμε όσον αφορά την κοινωνική τους κατάσταση, τις συντάξεις, τις προεπτικές στο σύγχρονο κόσμο εργασίας. Και αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Ότι όλοι λένε ότι βρίσκονται στο ίδιο σκάφο, αλλά κανεί δεν μπορεί να αναπτύξει τον δυναμισμό μέσω του οποίου μπορεί κανεί να νικήσει τα κύματα και να πλεύσει εν μέσω των απειλών και των κινδύνων σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί από την άλλη πλευρά κάθεται κάποιο σαν τον Πούτιν, ο οποίο δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τι δικέ μα ιδέε ελευθερία. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι από την άλλη υπάρχει και ο Τραμπ, ο οποίο δεν έχει ιδέα για την ε, δυνατότητά μα να οργανώσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη στην κοινωνία μας. Και τι περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν ε, μπορούμε να πυροδοτήσουμε αυτό το δυναμισμό ε, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ε, εμένα μου άρεσαν τα όσα είπε ο Πέντρο Σάντσεθ, γιατί εκπροσωπούν ένα πρόγραμμα ε, κοινή ε, καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υπόβαθρο των ανησυχιών που έχουν οι πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει να αντλήσουμε το δίδαγμα, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε αποτελέσματα. Ο Πέτρος Σάντσεθ ε, το εξέφρασε αυτό στην ομιλία του. Αυτό χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια της νέας εντολής. Και θα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μου άρεσε γιατί ε, αυτά υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας μιας ε, χώρας και θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπε ο Φραντ Τίμερμαντς, όπου η μοίρα της Ευρώπης ε, έχει, ε, συγκαθορίζεται. Μία χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ε, η οποία, μια χώρα η οποία γνωρίζει τις διαφορετικές ρίζες της. Μια χώρα όπου μπόρεσε να νικήσει το φασιστοειδές καθεστώς του Φράγκο μια χώρα που δεν θέλει να ξαναβυθιστεί στην εποχή της κατάργησης της δημοκρατίας και του ζώφου. Ε, στην Ισπανία και ξέρουμε ότι είναι σε καλά χέρια. Το πρόγραμμα το οποίο μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργό είναι πρόγραμμα το οποίο η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί ότι απηχεί τις αξίες της. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να μιλάμε πλέον για την οικονομία χωρίς την προεπτική της απασχόλησης των κατοίκων, των ε, πολιτών, αλλά δεν μπορούμε ε, να μην αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή παράλληλα η οποία θα σώσει τον πλανήτη. Αλλά αυτή η αλλαγή θα πετύχει μόνο εφόσον πάρουμε τους πολίτες με το μέρος μας. Μόνο εφόσον τους δώσουμε ελπίδες και προοπτικές. Δεν μπορεί να είναι μία αλλαγή η οποία να είναι εναντίον των πολιτικών. Δείτε την εμπειρία της Γαλλίας, την εμπειρία του Μακρόν. Πρέπει να ενισχύσουμε τους πολίτες ούτως ώστε να σταθούν στο πλευρό μας αυτή την αλλαγή. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική προοπτική, να της δώσουμε ένα αναθέσουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Ε, ναι, Βεβαίω ε, το διακύβημα είναι το πώς ε, γίνεται η διακυβέρνηση ε, και το μήνυμα από τη Μαδρίτη, το γεγονός ότι πετύχατε, Πέδρο Σάντσεθ, να φτιάξετε μια έξυπνη κυβέρνηση όπου πραγματικά μπορούν ε, υπουργοί με υψηλές δεξιότητες να συνενώσουν τις δυνάμεις της. Έχετε μια επίτροπο βιωσιμότητας και επιτέλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα όχι μόνο για την ισότητα των δύο φύλων αλλά ε, να ε, προωθήσετε γυναίκες με υψηλά προσόντα στην κυβέρνησή σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για το μέλλον της Ευρώπης και πολύ σωστά την ομιλία σας την συμπληρώσατε με τις ιδέες σας για το Brexit. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν σε ευχαρίστησε τους ε, Βρετανούς στρατιώτες που απελευθέρωσαν τη χώρα του από τους Ναζί. Εγώ είμαι Γερμανός, ο πατέρας μου ε, πέθανε στον πόλεμο, σκοτώθηκε στον πόλεμο και το ε, σπίτι μας βομβαρδίστηκε το 1943 και χάσαμε την μάχη της Βρετανίας. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, αλλά θα ε, λυπηθώ πάρα πολύ εάν χάσουμε τη μάχη που δίνουμε τώρα υπέρ της Βρετανίας. Το Brexit είναι μια κατάσταση από την οποία θα χάσουν ε, και η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι οικονομικά, πολιτικά και ηθικά ε, θα χάσουν. Οικονομικά διότι το Brexit θα αντιστοιχούσε ε, στο να αποχωρήσουν 19 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενιαία αγορά ταυτόχρονα. Πολιτικά, διότι, η, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα ήταν η φωνή της λογικής, ε, της επικουρικότητας, της αποκέντρωσης κλπ. Και ηθικά, διότι όπως είπαν προηγουμένως και πολύ σωστά διάφοροι ευρωβουλευτές, από το Brexit θα γίνουμε όλοι φτωχότεροι. Οι προηγούμενες συζητήσεις δείξαν ότι σχεδόν όλοι ε, λυπούνται για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτό από του ανθρώπου που βρίσκονται εδώ στα αριστερά μου, αλλά ούτε ένα δεν έχει προσφέρει μια λύση για να σταματήσει το Brexit και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Ε, πάνω από 140 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου απευθύνθηκαν ε, στον ε, λαό της Βρετανίας, ε, τους ζητάνε δεύτερο δημοψήφισμα. Σύμφωνο με αυτό, αλλά θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει νωρίτερα, διότι σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Φερχόφστατ, δεν είναι το πρόβλημα μόνο οι διαμάχες εντός ε, του συντηρητικού κόμματος. Υπήρχαν ε, λόγοι που το Ηνωμένο Βασιλιά άρχισε να σκέφτεται την Ευρώπη. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, μιλούσαμε για την επικουρικότητα, αλλά τι έγινε συγκέντρωση της εξουσίας. Μιλούσαμε για ανταγωνισμό, βλέπουμε όμως όλο και περισσότερη εναρμόνιση. Μιλούσαμε στη συνθήκη της Λισαβόνας για την ευθύνη κάθε κράτους για το χρέος του, αλλά τελικά τι κάνουμε, κοινωνικοποιούμε το ε, χρέος. Ήρθε η ώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αρχίσουν να κάνουν ε, άλλα πράγματα. Αναφέρθηκε μια νέα συμφωνία ώστε η ΜΕΗ να συγκεντρώσει την πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου της. Αλλά ας ε, κάνουμε κάτι άλλο. Ας δώσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια ε, συμφωνία που ε, θα, την, που θα το κάνει να θέλει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε ότι έχουμε ευθύνη για το Brexit. Ας προσφέρουμε λοιπόν μια νέα συμφωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να παραμείνει εντός του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί μόνο να είναι μια ειδική ε, προσωρινή συμφωνία για τη μετανάστευση. Αντί πάντα να κατηγορούμε τη Βρετανία, ας αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και οι Βρυξέλλες αποτελούν μέρος του προβλήματος. Θα πρέπει να γίνουμε όμως μέρος της λύσης. Ας ε, αγωνιστούμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο των Φιλελευθέρων, ο κύριο Φερχόφστατ. Μάλιστα, τέσσερα λεπτά, γιατί έχω έναν Ισπανό, έναν Καταλανό και έναν Βάσκο συνάδελφο που θέλουν να πάρουν το λόγο μετά από μένα και τη θέλω τη ζωούλα μου ακόμη. Ε, Ένα χαρακτηριστικό της Ισπανίας ε, και εσείς είστε ζωντανή απόδειξη αυτού είναι πως ίσως είστε η, πιο ε, φιλοευρωπαϊκή χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή γιατί έχει το θάρρος να μιλά για ομοσπονδιακή Ευρώπη. Πολλοί από τους συνάδελφούς σας που ήρθαν εδώ δεν είχαν αυτό το θάρρος. Δεν είναι τυχαίο πιστεύω αυτό. Πιστεύω διότι η ευρωπαϊκή ιστορία και η ισπανική δημοκρατία είναι αλληλένδετε Πιστεύω επίσης επειδή τα τις τελευταίες δεκαετίες ε, το Υπουργείο Εξωτερικών σας ε, και μέλη εδώ σε αυτήν την, ε, την, την η ο Μέντες Δεβίγκο, η Παλάσιο ο Μιγγέλ Μορατίνος που ήταν πρώην ε, υπάλληλο και τέλος ε, υπάρχει ανταγωνισμός στην ισπανική πολιτική ώστε να, ποιος θα είναι ο πιο φιλοευρωπαϊστής από τα κόμματά σας ανάμεσα στο ΠΠ, το ΨΟΕ και τους ε, Σιουταδάνους και πολύ μου αρέσει αυτό να βλέπω και θα ήθελα σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει αυτό το είδος η άμυλα ποιος θα είναι ο πιο φιλοευρωπαϊστής δηλαδή ανάμεσα στα κόμματα. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν ξέρω, είναι η 15η συζήτηση που κάνουμε για το μέλλον της ε- Ένωσης και λίγο αισθάνομαι μια... Έχω μπερδευτεί γιατί κάθε φορά έρχεται ένας πρόεδρος, έρχεται ένας πρωθυπουργό, κάνει ένα ολόκληρο κατάλογο των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών που πρέπει να κάνουμε, κοινωνική πολιτική, φορολογική πολιτική, μεταναστευτική πολιτική, ευρωπαϊκό στρατός και ποτέ δεν λέμε γιατί δεν το κάνουμε στην πράξη. Ποιο είναι το εμπόδιο. Γιατί πάντοτε ενεργούμε πολύ λίγο και πολύ αργά σε σύγκριση με τους Αμερικανούς, ας πούμε, που σε 9 μήνες ε, ε, τα κατάφεραμε την κρίση και εμείς μετά από 9 χρόνια δεν έχουμε ακόμα τραπεζική ένωση. Τεράστια τραγωδία στη Μεσόγειο και σας συγχαίρω ε, ε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τους πρόσφυγες του Ακουάριου. Αλλά ας είμαστε ειλικρινεί, αυτή είναι η συνέπεια ε, της απάνθρωπης ε, νασιοναλιστικής, εθνικιστικής δηλαδή πολιτικής του Σαλβίνη. Ε, και είναι και λόγω της έλλειψης ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί δεν έχουμε ακόμα τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί ακόμα δεν έχουμε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, για παράδειγμα, μετά από τόσο πολλά χρόνια τραγωδιών στην Μεσόγειο. Γιατί δεν έχουμε ευρωπαϊκό στρατό ήδη σήμερα, γιατί ακόμα αγωνιζόμαστε με τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, εννέα χρόνια μετά από την αρχή της κρίσης. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για μένα και ελπίζω ότι στην απάντησή σας σε λίγα λεπτά θα μας μιλήσετε για αυτό το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κακούς θεσμούς αυτή τη στιγμή στην Ένωση και οι καλοί θεσμοί οδηγούν σε κακά αποτελέσματα. Ενώ οι καλοί θεσμοί καλά αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι και θέλω να το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια μαζί με κάποιου από εσά. Είναι ο κανόνα τη Ομοφωνία που ισχύει στην Ένωση και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η έλλειψη ισορροπία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποφασίζει με την πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εξακολουθεί να αποφασίζει